a las explicaciones de voto. Εξηγήσεις ψήφου. Πρώτος, όσον αφορά την έκθεση Μωράες, ο κύριος Μαστέλα. Τέλα νοστά Δεν είναι εδώ. Κύριος Χάναν, λοιπόν. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο. Αισθάνομαι ότι μπήκα σε κάποια τρύπα του χωροχρονικού συνεχούς και γύρισα στην ε, δεκαετία του 70 σε έναν κόσμο βιομηχανίας που λέγεται το κράτος, ε, πολιτικών εισοδηματικών, τιμολογικών, επιδοτήσεων σε μη, κερδοσκο... επιχειρήσει. επιχειρήσεις. Θα μπορούσα να διαβάσω τον κατάλληλο ψηφοφορίων που ψηφίσαμε. Επιδοτήσεις ε, Σαϊαμούρα στην, στη Χαϊδελβέργη, στην AGE στην Γερμανία, Βικερπόλσκι Οτομοτίβ στην Πολωνία, στην Aragon Retail στην Ισπανία, Κομμουνιτάδ Βαλενσιάνα και στη Χριστιφαντουργικά, ε, για τις λίθους στην ε, Βαλενσιάνα, στην Ετσεγεύσκη Ποσνάν στην Πολωνία και λοιπά. Τη δεκαετία του 70 μιλούσαμε για την επιλογή νικητών. Εδώ επιλέγουμε ιτρουμένους. Και εδώ έχει αποτύχει ελεύθερη αγορά, έχουν αποτύχει γιατί το κάνουμε, γιατί είναι ένας μηχανισμός για κατανομή πλούτου σε ευνοούμενε ομάδε πελατών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, αυτή αυτά είναι ανόητα. Ήσασταν πάρα πολύ επιτυχεί ηγέτη δυτικών στην Καταλωνία. Ξέρετε πόσο είναι σημαντικό να είναι ελεύθεροι λαοί και οι αγορέ. Το ίδιο και οι ψηφοφόροι μα. Τα χρήματα τελειώνουν και φτάσαμε στη στιγμή όπου, όπω έλεγε ο Τζορτ Όρουελ, οι λαοί θα αποτινάξουν το σύστημα όπω ο άλογο αποτινάσει τα Ευχαριστώ. Έκθεση Γκρίσμπεκ. Έχει το λόγο η κυρία Μορκονάιτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ότι έχει ισχυρή θέση. Έκανε ένα βήμα προς τη συνεργασία στο Νότιο Κάφκασο. Ο Νότιος Κάφκασος και η Γεωργία έχουν στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μου, η Λιθουανία, πάντα έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Γεωργία. Υποστηρίξαμε σε δύσκολες στιγμές αυτή τη χώρα και όχι μόνο σε επίπεδο κρατικό. Η κοινωνία μας είχε εκφράσει μεγάλη υποστήριξη προς την χώρα αυτή. Ελπίζω ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει η Γεωργία να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτή η χώρα καταβάλει πολλές προσπάθειες να μετάσχει στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσουμε. Η διευκόλυνση θεωρήσεων διαβατηρίων θα διευκολύνει την κινητικότητα των ανθρώπων, θα βελτιώσει την συνεργασία και ανταλλαγή εμπορική και πολιτισμική. Συγχαίρω το λαό της Γεωργίας για την απόφαση που ελήφθη. Μάλλον χαίρομαι την απόφαση που ελήφθη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στείλαμε ένα μήνυμα ότι είναι ευπρόσδεκτοι στην Ευρώπη οι, οι, Γεωργιανοί. Περνάμε στην έκθεση Μανέσκου τώρα. Ο κύριος Καλινιόφσκι έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε Τώρα τέτοια ποσά, τεράστια ποσά, να πάνε χαμένα. Και γι' αυτό πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση των κονδυλίων, ο τρόπος απορρόφησής τους. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν το πιο σημαντικό ρόλο. Καλό θα είναι να εξεταστεί η διασυνοριακή συνεργασία να εξασφαλιστούν απλουστευμένες διαδικασίες, να χορηγηθούν περισσότερα κονδύλια για την εκπαίδευση στα επιμέρου κρατη κράτη-μέλη και να υποστηριχθεί ο εξυγχρονισμό και η ανάπτυξη των συστημάτων τη κοινωνική πληροφορία. έτσι ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Πρίλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Μια διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα, η καλύτερη συμμετοχή των υπερεθνικών αρχών για τον καθορισμό των αναπτυξιακών πολιτικών, κυρίως στον τομέα της σύγκλησης. Πρέπει να αυξηθεί η δυνατότητά τους να κινηθούν σε επίπεδο κρατών μελών και να συμβάλλουν στην λειτουργία της όλης αγοράς για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην, για την ανάπτυξη θα πρέπει να γνωρίζει κανείς σε, τοπικό επίπεδο τις ανάγκες περιφέρειας. Γι' αυτό έχουμε τη σχέση μεταξύ της εδαφικής συνοχής και της πολυεπίπεδης προσέγγισης. Χρειαζόμαστε πιο ευέλικτη προσέγγιση. Μείωση γραφειοκρατίας. Επιτάχυνση. Ποιότητα επενδύσεων για την ανάπτυξη των περιφερειών μεγαλύτερη βοήθεια προς τις αρχές που χειρίζονται τα ποσά από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μείωνε τα σφάλματα που διαπιστώσαμε στο παρελθόν σε αφορά τους ελέγχους πρώτου επίπεδου. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πυρίλο. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μεσάρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η περιφερειακή πολιτική πρέπει να είναι και δυνατόν να ελεγχθεί και να δρά αποτελεσματικά για να είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον στους Ευρωπαίους πολίτες και υποστηρίζω την ε, πρόταση διότι βλέπω ότι η πιο στενή περιφερειακή συνεργασία θα βελτιώσει το επίπεδο όλων των κρατών μελών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να απευθυνθούμε προς τους συμπολίτε μας και να τους καλέσουμε να εποφεληθούν αυτής της υπερσυνοριακής συνεργασίας. Θα πρέπει να συμπράξουν ο το δημόσιο τομέα, να ενώσουν τα χέρια και να αναλάβουν δράση προκειμένου να υποστηρίξουν και να βελτιώσουν το επίπεδο ευημερία προ των πολιτών. Οι τοπικές περιφερειακές αρχές έχουν και πολύ μεγάλο, επίπεδο, πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού αυτό αποτελεί παράγοντα και αβεβαιότητας αλλά και ε, ε αισιοδοξία. Και νομίζω θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Κύριο Στάκουλα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την κυρία Μανέσκου την εισηγήτρια για την εξαιρετική της έκθεση που είναι τόσο σημαντική για την περιφερειακή πολιτική και για την καλύτερη διαχείριση. Η καλύτερη διαχείριση, governance, ε, βασίζεται στο, στην αρχή της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης. Δεν μπορούμε να διαλέγουμε μόνο το καλύτερο κομμάτι της τούρτας, πρέπει όλα τα εργαλεία της περιφερειακής πολιτικής να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσει αυτή να υλοποιηθεί. Όταν διαβάζουμε τα κριτήρια, όταν απαριθμούμε τα κριτήρια, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε σε ορισμένες μόνο χώρες, γιατί αυτό δεν είναι βιώσιμο κριτήριο. Οι χώρες, οι αραιοκατοικημένες περιοχές πρέπει επίση να τύχουν μιας καλής διακυβέρνησης και διαχείρισης, κύριε Πρόεδρε, εφόσον μιλάμε για ισότιμη τη αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Τακούλα. Τώρα η έκθεση Δίας Δεμέρα, πάλι ο κύριος Τακούλας. Κύριε Πρόεδρε, τα θέματα της μετανάστευσης αυτή τη στιγμή είναι επίκαιρα για όλη την Ένωση και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα δίκτυο όπως ζητήσαμε στην έκθεση αυτή και η Ένωση να μπορέσει να εφαρμόζει ίση και δίκαια μεταχείριση των μεταναστών. Δυστυχώς υπήρξαν παραδείγματα της τέτοιας μεταχείρισης. Υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν και καταστάθηκαν στην Ευρώπη αλλά δεν δέχονται τις βασικές τις αρχές. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ώστε οι βασικές αρχές τις οποίες στηρίζεται η Ένωση να εφαρμόζονται από όλους. Πρόκειται για θέμα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, κτλ. Όλα αυτά είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, τα θεωρούμε ζωτικά <coughs> και γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθεί και η δεοντολογική βάση στην οποία θέλουμε να εφαρμόζουμε και εμείς την μεταναστευτική μας πολιτική και οι μετανάστε την διαβίωση του στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κύριε Τακούλα για την έκθεση Ματιού. Για την έκθεση λέω Ματιού, ο κύριος Αντώνιο Τσιγραπτός, κυρία Βέρμαν Γραπτός. Για την έκθεση Χιμένες, ποιος είπε ο κύριος Ρούντι απουσιάζει, Αντωνιώτσι Γραπτός. Ματσέσκο, η κυρία Τσέσκοβα μάλλον. Μια Τσέσκοβα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να είχα λάβει το λόγο πριν από την ψηφοφορία γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το εργαλείο αυτό γιατί εδώ διώκονται γυναίκες και χρειάζονται προστασίας Λυπούμε λοιπόν ιδιαίτερα γιατί το κείμενο που εγκρίναμε σήμερα δεν βασίζεται σε σταθερή σωσταθρό νομικό υπόβαθρο. Ίσως μπορεί να βελτιωθεί ακόμη για να το εκμεταλλευτούμε όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό και εγώ απέσχομαι. Ρόντι. Με συγχωρείτε, σας έψαχνα, αλλά αλλού δεν σας είχα δει εδώ, λοιπόν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δυστυχώ, δεν λειτουργήσε το μηχάνημά μου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορία. Θα είχα όμως εγκρίνει, διότι πρόκειται για πολύ σημαντικό θέμα και έπρεπε το Κοινοβούλιο να εγκρίνει γιατί η νομοθεσία αυτή είναι ουσιώδης και η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων είναι κάτι το πολύ βασικό για να δημιουργηθεί ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας δικαιοσύνης κλπ. ε, αυτή τη στιγμή δίνεται ένα νομικό υπόβαθρο ώστε να μπορεί ένα κράτος μέλος να εφαρμόσει μια δικαστική απόφαση που ελήφθη σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό αφορά ιδιαίτερα το θέμα της βίας κατά των γυναικών και άλλων. Έτσι ώστε να μπορέσουν τα θύματα να αποφασίσουν να παραμείνουν οπουδήποτε θέλουν μέσα στην Ένωση και να τύχουν της ίδιας προστασίας. Ευχαριστώ έκθεση Bauer, ο κύριος Αντωνιώτης Γραπτός, κυρία Ντότς. Ντότς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, η πορεία ανθρώπων είναι σοβαρότατο ζήτημα. Από το 2008 35 άνθρωποι διασώθηκαν από την εκμετάλλευση στην εκλογική μου περιφέρεια της Βορείου Ιρλανδίας. 25 από αυτούς διασώθησαν το 2009. Όμως ουδής κατεδικάστη για αδίκημα που σχετίζεται με την εμπορία ανθρώπων είναι σύγχρονη μορφής δουλεία σοβαρό έγκλημα και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου. Πολλές γυναίκες που διεσώθησαν στην Βόρεια Ιρλανδία είναι από την Άπο Ανατολή και μέσω συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος που κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα και εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους και για εργασία και σεξουαλική εκμετάλλευση. Γι' αυτό βρήκα σε αυτή τη θέση. Υπάρχουν πολλέ ε, ε πολύτιμε στοιχεία στην έκθεση και είναι ένα τομέα που μπορεί να επιτευχθεί συνεργασία μεταξύ εθνικών αστυνομικών δυνάμεων και η αστυνομική δύναμη τη Βορείου Ιρλανδία έχει ηγηθεί στο θέμα. Παρ' όλα αυτά, είχα απόσχεια από την ψηφοφορία, διότι πιστεύω ένθερμα ότι ο καθορισμός ελάχιστων ε, ε, ε ποινών είναι κάτι που αφορά τα κράτη-μέλη και μόνο. Ευχαριστώ. Ο κ. Τακούλα έχει το λόγο και πάλι. Ε, κύριε Πρόεδρε, όταν μιλάμε για εμπορία ανθρώπων, είναι τα σοβαρότερα ζητήματα. Η μεγαλύτερη απειλή που γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωριστεί αυτό, να αναγνωρίσουμε τη σοβαρότητά του, ακόμα και αν συχνά σκριβόμεθα πίσω από αυταπάτες ότι έχουν επιληθεί αυτά τα προβλήματα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει ο καθένας να απολαμβάνει τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Στα αγγλικά μιλάμε για human trafficking. Τίποτα ανθρώπινο δεν υπάρχει σε αυτήν την ε, δραστηριότητα. Είναι κάτι φρικτό. Στερούμε από τους ανθρώπους την αξιοπρέπειά τους, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και οι ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Η πορνεία, το εμπόριο οργάνων, για μεταμοσχεύσεις είναι η βασική στόχη αυτού του εμπορίου. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να κινηθεί, να πάψει να μιλά και να δράσει ούτω ώστε στην επικά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να τεθεί τέρμα οριστικά στο εμπόριο ανθρώπων. Θα πρέπει να επιβληθούν αποτρεπτικέ κυρώσει, ούτω ο καθένα να μπορεί να ζει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ κύριε Τακούλα. Η κυρία Ζαμπόρσκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Υποστήριξα την οδηγία γιατί θεώρησα ότι το εμπόριο ανθρώπων στερεί από τον κόσμο την ελευθερία του. Χαίρομαι που βλέπω ότι αυτή η οδηγία καθορίζει κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν οι χώρες, που πρέπει να ενισχύσουν οι χώρες την νομοθεσία τους, να την κάνουν αυστηρότερη. Οποιοδήποτε είδος εμπορίου χρειάζεται και τον αγοραστή. Πολύ συχνά αυτοί που αγοράζουν είναι πλούσιοι από δημοκρατικέ χώρε. Μπορεί να είναι και ο γείτονά μα που αγοράζει. Ε, η έκθεση επίσης ε, αναφέρεται στα θύματα, αλλά θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να προσέχουμε και οι ευάλωτοι ε, να προστατεύονται, τους βοηθήσουμε να προστατευτούν, να μην γίνουν θύματα. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους νέους, δασκάλους στα σχολεία, γιατί πρέπει να ενισχύσουμε τον τομέα της πρόληψης. Και αυτό είναι κάτι που σχετίζεται και με τη ζήτηση βέβαια. Ευχαριστώ κυρία Ζαμπόρσκα. Έκθεση Γκρίσμπεκ τώρα. Η κυρία Ροντζούλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πήρα το λόγο για το εμπόριο των, ανθρωπίνων δικαιω... Ε, των ανθρώπων ήθελα να μιλήσω. Το εμπόριο ανθρώπων. Ζήτησα το λόγο όσον αφορά τη ε, δήλωση ψήφου για το εμπόριο ανθρώπων. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Όχι επανειστοχή των ε, εκείνων που διαμένουν παράνομα σε κάποια χώρα. Δεν θέλετε να μιλήσετε για αυτό το θέμα. Ε? Λυπάμαι. Θα σας δώσω το λόγο για να κάνετε επεξήγηση ψήφου όσον αφορά την έκθεση Bauer. Ευχαριστώ Πρόεδρε ψήφισα προφανώς υπέρ της εκθέσεως Μπάουερ διότι η καταπολέμηση των ανθρώπων είναι και πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητά μας. Αυτό το φαινόμενο πήρε τέτοιες αναλογίες που μπορεί να θεωρηθεί νέα μορφή σκλαβιάς νέα μορφή δουλεία. Η πιο ευάλωτη τη κοινωνία, οι γυναίκε, τα παιδιά μεταφέρονται σε άλλε χώρε και αποτελούν κείμενο εκμετέλευση μέσω των χειροτέρων μορφών πορνεία, δουλεία και πορνογραφία. Αυτό το φαινόμενο κάθε χρόνο αφορά εκατομμύρια θύματα σε όλο τον κόσμο. 500.000 θύματα μόνο στην Ευρώπη. Ποιο αυτό που εκμετάβεται αυτό το φαινόμενο είναι τα εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποίησαν εμπορεύματα του ανθρώπου για τα κέρδη του. Όπως υπογραμμίζεται από την έκθεση θα πρέπει να εφαρμοστούν δράσεις στι χώρες καταγωγής και τι οποίε μεταφέρονται τα θύματα αυτού του εμπορίου. Η λύση θα μπορούσε να εξευρεθεί μόνο μέσω μιας κοινή προσπαθία που σημαίνει προσπάθεια ευαισθητοποίησεως συλλογική και σημαίνει υποστήριξη των θυμάτων, βοήθεια για τα θύματα και πάνω απ' όλα καταπολέμηση των βασικών αιτίων του φαινομένου, ούτω ώστε να βοηθήσουμε τι χώρε που εμπλέκονται να αναπτύξουν επαρκή νομοθεσία, ούτω ώστε να αντισταθούν σε κάθε μορφή σκλαβιά. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντέβα. Για ποια έκθεση θα μιλήσετε. Για ποια. Εκτός μικροφώνου ο κ. Ντέβα, οι διερμηνεί δεν μπορούν να τον ακούσουν. Α, έκθεση Γκρίσμπεκ, λέει ο Πρόεδρος. Καλώς. Μάλιστα. Καλώς. Πάμε στην έκθεση Γκρίσμπεκ, λοιπόν. Και το λόγο δίνω εν πρώτης στον κύριο Γιάρ και μετά στον κύριο Ντέβα. Ο κύριος Γιάρ, έχετε το λόγο για την έκθεση Γκρίσμπεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που εδώ στο Κοινοβούλιο μπορέσαμε να ρυθμίσουμε και το ζήτημα της συμφωνίας με τη Γεωργία αλλά και εκείνο της ε, συμφωνίας για την ε, επαναπροώθηση ατόμων που δεν είχαν κατάλληλη άδεια παραμονής. Το λέω αυτό κατά αυτόν τον τρόπο για να σημειώσω ότι είναι καλό να ασχολούμαστε και με τα ευχάριστα ζητήματα, με τα θετικά, αλλά και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Και ελπίζω ότι θα έχουμε σύντομα, σε ένα χρόνο, την επόμενη διάμεση έκθεση για να δούμε πώς εφαρμόζεται αυτή η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας, τι δύο αντίκτυπο είχε και ελπίζω την επόμενη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να συζητήσει πιο εντατικά ε, και να λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις ε, για την υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δίβα έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί η ομάδα μου και εγώ δηλώσαμε αποχή στο θέμα της, ε, των δυνατοτήτων δοχές αντίδρασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δει ότι είναι όλο και πιο ε, υψηλά τα, ε, υψηλές προσδοκίες ως προς την ταχεία αντίδραση των ομάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο. Και ναι, μεν θεωρώ ότι υπάρχει, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ να θεσπιστεί μια νέα ομάδα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, βεβαίως θα πρέπει με την ευρύτερη αναπτυξιακή κοινότητα να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τέτοιες εξελίξεις μπορούν να λαμβάνουν χώρα μόνο εντός των υφισταμένων μηχανισμών και δομών, όπως ε, των κοινοτικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Γιατί λοιπόν χρειάζεται κάτι διαφορετικό για τις ανθρωπιστικές ε, καταστροφές. Γιατί να είμαστε μόνο εμείς εκείνοι οι οποίοι ανταποκρινόμαστε θα έπρεπε να βελτιώνουμε και την ανταπόκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να ενισχύουμε τη δυνατότητα ανταπόκριση των αντισωμένων χωρών, των περιφερειών του, των υποπεριφερειών στι πληττόμενε περιοχέ, έτσι ώστε μαζί με αυτέ, μαζί με τη διεθνή κοινότητα να αναλαμβάνουμε τη σχετική δράση. Διαφορετικά, όλη τη σκληρή δουλειά θα την κάνουμε εμεί και οι άλλοι απλώ θα επαναπαύονται. Ευχαριστώ πολύ, Λίγο Πρόεδρο. Κύριε Ντίβα, πρέπει να σας πω ότι δεν θα έπρεπε κανονικά να προβείτε σε επεξήγηση ψήφου, διότι δεν έγινε συζήτηση για το θέμα. Αλλά τώρα έγινε. Μπράβο σας. Εν τέλει, έκθεση Λούαν. Κύριος Καλινόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλοί είναι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγνοούν την σημασία της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη των περιφερειών και των κρατών μελών. Η πολιτική αυτή στηρίζεται σε μια βασική ιδέα να εξασφαλίσει πρόσβαση στις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη σε βασικές υποδομές, ενέργεια, και άλλους σπόρους Και έτσι, για αυτό το λόγο έχει τόσο μεγάλη σημασία η συνοχή. Πρέπει λοιπόν να συντονίσουμε τις προσπαθίες μας και να εξασφαλίσουμε καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων. Επιπλέον δε, Ξέρουμε πολύ καλά ότι η πολιτική συνοχή έχει αντίκτυπο πολύ πιο ξεκάθαρο στι τοπικέ κοινωνίε και γι' αυτό θα πρέπει να, αυτή, να υποστηρίξουμε αυτή την ιδέα. Κύριο Νικολάτσικ, παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνουμε επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Λουχάν, τελευταίο θέμα στις προφορίες μας. Το ζήτημα της συνοχής σημαίνει υποστήριξη προς τις περιφέρειες. Η ανταγωνιστικότητα όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η συγχρηματοδότηση από τα διευθυντικά ταμεία έχει αποδειχθεί πολύ ικανοποιητική μέθοδος και έχει εξασφαλίσει βελτίωση των υποδομών που αποτελεί πολύ σοβαρό στόχο διότι υπάρχουν πολλές περιφέρειες που χρειάζονται ανάπτυξη των υποδομών τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την οικονομική εφημερία. Η κοινωνική συλλογή επίση επεδείχθη χρήσιμο εργαλείο και σε περίοδο οικονομική κρίση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειε αυτή, Επίση, η οικονομική ανταγωνιστικότητα των περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε ότι σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο τη ανεργία και ιδιαίτερα με την ε, ύπαρξη και απασχόληση καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού. Η κοινωνική συνοχή αποτελεί σημείο κλειδί για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο επίσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μικολάσιτς. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της συνεδρίασής μας και διακόπτουμε μέχρι τις, 5, μέχρι τις 3 το απόγευμα που θα ε, συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ.